Good morning, dear colleagues. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε λοιπόν με την ε, έγκριση της σημερινής διάταξης. Το σημείο 21 θα εξεταστεί μετά το σημείο 23. Το δε σημείο 2 θα εξεταστεί μετά το σημείο 17. Και το 16 και το 21 αναβάλλονται. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει και αν δεν λάβουμε καμία αντίρρηση μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση, θεωρείται ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη 24η Ιανουαρίου και τη 21η και 22η Φεβρουαρίου εγκρίνονται. Α περάσουμε στο σημείο 4. Αντικατάσταση του παραρτήματο α του κανονισμού 848 του 2015 περί των διαδικασιών εφαρεγγιότητας. Ο κύριος Ταντέους Ζεύσκα είναι ο εισηγητής για το σημείο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Ζεύσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, για άλλη μία φορά γίνεται το ερώτημα ε, αυτό θα ε, ήθελα να ασχοληθώ με τα ερωτήματα τα οποία αφορούν την όλη ε, διαδικασία από την ε, αρχή της ε, νομοθετικής περίοδου ε, είχαμε ε, επιτυχημένες διαπραγματεύσεις ε, με το Συμβούλιο και επίσης εισάγαμε τον κανονισμό από το 2014. Από τον Ιούνιο του 2016 λοιπόν ισχύει ο συγκεκριμένος κανονισμός ε, και συγκεκριμένα το κομμάτι το οποίο αφορά την ε, δικτύωση των ε, μητρώων αφαιρεγγιότητας και αυτό θα τεθεί σε ισχύ από το 2019. Ε, η όλη διαδικασία είναι ε, ιδιαίτερα δυναμική ε, και κάθε κράτος μέλος προσπαθεί να προσαρμόσει τους νόμους του πάνω σε αυτό. Για σκέφτεται το καλό των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων σκεφτόμουν να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις στη διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Ε, ε, το σημαντικότερο θέμα είναι τα κοινωνικά ζητήματα, τα οικονομικά ζητήματα ε, πάντοτε εμφανίζονται νέες λύσεις που αρχίζουν να ισχύουν στην ε, στο συγκεκριμένο κανονισμό. κανονισμό. Έχουμε ε, δύο παραρτήματα. Στο, στο Α έχουμε τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητες, ενώ στο Β έχουμε την περιγραφή των οργάνων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της διαδικασίας ε, επειδή λοιπόν σε ε, διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν κάποιες αλλαγές θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς ε, αυτές τις, αυτές, αυτές τις αλλαγές μέσω μιας κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Το είχαμε ε, στην αρχή αυτό το 2016 όταν στο πολωνικό ε, δίκαιο υπήρξαν κάποιες ε, αλλαγές και έπρεπε να γίνει η προσαρμογή. Πλέον έχουμε το νέο αίτημα από Κροατία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Λετωνία καθώς επίσης και το Βέλγιο, στρέφονται λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροπολογίες για να γίνουν οι απαραίτητες ε, προσαρμογές, ε, διότι στον κανονισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες διαδικασίες, οι αλλαγές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν που έγιναν στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αξιολόγησει ήδη το συγκεκριμένο θέμα ε, και ότι θα μας παράσχει τις ε, πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες της, διότι θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο, εργαζόμαστε παράλληλα, δεν περιμένει ο ένας τον άλλον το πρόβλημα λοιπόν είναι ε, τεχνικό ε, και ελπίζω ότι και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη θα αξιολογήσουν, έχουν κάνει ήδη μια αξιολόγηση των εργαλειών τους ε, και ότι όλη η διαδικασία θα ολοκληρωθεί γρήγορα. Και αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει πράξει ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίσκα. Ε, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στα ε, μέλη που θέλουν να κάνουν κάποια σχόλια. Όχι. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν ε, σχόλια, θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Κομισιόν ή η Προεδρία του Συμβουλίου θα ήθελαν το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι στηρίζουμε την έκθεση του εισηγητή και επίσης επιβεβαιώνουμε την συμφωνία μας για τις τροπολογίες που ετέθησαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Να δώσω απλώς κάποιες σύντομες εξηγήσει σε σχέση με τα όσα ήδη είπε ο εισηγητής. Οι τεχνικές τροπολογίες οι οποίες προτείνονται στο πρώτο παράρτημα του κανονισμού διαδικασιών εφερεγκαιότητας περιλαμβάνονται νέες εθνικές διαδικασίες εφερεγκαιότητας, οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί στις διάφορες εθνικές νομοθεσίες. Κατά τη διάρκεια των συστήσεων που γίνανε στο Συμβούλιο, πολλά κράτη-μέλη επικαιροποίησαν την εθνική τους νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως πολύ προσεκτικά εξέτασε τη συμμόρφωση των εθνικών αυτών νομοθεσιών και κοινοποίησε στα κράτη-μέλη ποιε είναι οι απαιτήσει του κανονισμού διαδικασιών εφερεγγιότητα. Μετά την αξιολόγηση αυτή, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ε, οι απαιτήσει του κανονισμού ε, πληρούνται και συνεπώ επιβεβαιώνουμε ότι όντω συμφωνούμε με το κείμενο του Συμβουλίου και τονίζουμε ότι όντω ε, οι τροπολογίε αυτέ, οι τροποποίησει αυτέ είναι τεχνική φύσεω και πρόκειται για μια τεχνική αξιολόγηση που γίνεται και πληρούνται σε κάθε περίπτωση προποθέσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Um, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιέσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε την Κομισιόν για την ε, δήλωση που έκανε. Και σας προτείνω το εξής, αυτή τη διαδικασία λοιπόν για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 1η ε, Απριλίου. Εάν δεν υπάρχουν τροπολογίες ή αν δεν είναι πολύ περίπλοκες αυτές οι τροπολογίες, τότε στην επόμενη συνεδρία της Νομικής Επιτροπής ε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε και να ψηφίσουμε το κείμενο αυτό. Και αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σβέσκα. Ναι, θυμάμαι κι εγώ ότι η 11η Απριλίου είναι η ε, προθεσμία και θα δούμε πότε θα γίνει η ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5 που αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση πρόκληση στους τομείς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αστικής ευθύνης. Η κυρία Ζωέλ Μπερζερόν είναι η συγγήτρια και θα της δώσω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ κυρία Μπερζερόν. Ευχαριστώ Λάουρα, ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τη συμβολή που είχατε ε, σε αυτήν την έκθεση που αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση. Έχουν ε, κατατεθεί 149 τροπολογίες που καταδεικνύουν το ενδιαφέρον σας, ε, για το οποίο σας ευχαριστώ. Σας προτείνω να ξαναδούμε κάποιες από αυτές τις τροπολογίες έτσι ώστε να τις ε, συζητήσουμε. Επίσης υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία δεν πολύ κατανόησα γιατί ενδεχομένως η μετάφραση δεν είναι πολύ ποιοτική. Ε, πολλές τροπολογίες στην ιδεολογική σκέψη 1, ε, γιατί πολλοί εισηγητές, οι συνεισηγητές τουλάχιστον ε, οι έχουν υποβάλει τροπολογίες, γιατί θεωρούν ότι δεν συμφωνείται με την άποψη ότι είναι περιθωριακό το, η αγορά της Εκτύπωση της τρισδιάστατης εγώ θεωρώ ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, μαζί με τους ε, οι υπευθύνους και τους εμπορευμένους του τομέα να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Ε, υπάρχουν λοιπόν οι τροπολογίες Δεγράντες Pascual, Μπιογκά και Καρίμα ε, καθώς επίσης οι τροπολογίες οι οποίες προσθέτουν κάποια ε, χρήσιμα στοιχεία, ε, όπως αυτή του κυρίου Μπούντα, ο είναι πάντα πολύ σαφής όσον αφορά το γάμα σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουν στις διάφορες, στους τομείς δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να έχουμε ε, τροπολογία συμβιβαστική, γιατί οι τροπολογίες 25 και 27 στοχεύουν στο ίδιο σημείο, δηλαδή να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι ε, πολλοί είναι οι τομείς αυτοί οι οποίοι ε, τους οποίους αφορά η τρισδιάστατη εκτύπωση. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά εγώ πιστεύω ότι η ιατρική, η αεροναυτική, η αεροδυναμική διαστημική, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι κατασκευές, η αρχιτεκτονική, η αρχαιολογία επίσης, το design ε, είναι η πρώτη... Ε, Τομεί που μου έρχονται στο μυαλό. Συμφωνώ με τον κύριο Τεγκράντες Πασκουάλη όταν λέει στην τροπολογία του 31 ότι ε, η απομείωση τη διάσταση εκτύπωση σε ε, ε, πολύ σημαντικού τομεί, όπω είναι η αεροναυτική ή η ιατρική θα πρέπει να ειδωθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα δώσει καινούργιες εκτυπωση θα δωσει καινούργιε δυνατότητε στην έρευνα και την ανάπτυξη χρησιμοποιώντα ή εφευρίσκοντα Νέε τεχνολογίε Όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη ε σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση που μπορεί να είναι λιγότερο επαχθής και λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία, ε, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να βρούμε μία έναν συμβιβασμό ε, με τις τροπολογίες 37, 38, 39, 40, Χρυσόγονου, Μασταλκά, Γουγκά, ε, του κυρίου Λεμπρετών και της κυρίας Μπουτενέ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι αντίθετα από την ανησυχία που δείχνουν ορισμένοι μεταξύ ημών, ε, η εκτί, τριδιάστητη εκτύπωση δεν είναι ε, πάντα ε, παράνομη και δεν προκαλεί πάντα πλαστογράφηση. Η Μαστάλκια και θρυσόγονος καθώς επίσης και ο Λεμπρετών που ανέφερα προηγουμένως και της κυρίας Μπουτενέ νομίζω ότι μπορούν να ολοκληρώσουν συμπληρώσουν πολύ θετικά τη δικιά μου σκέψη. Αγαπητέ συνάδελφε, Υπάρχει μια ε, τροπολογία σας ε, που δεν έχω κατανοήσει, είτε εγώ έχω πολύ στραβό κεφάλι, είτε η μετάφραση δεν είναι πάρα πολύ καλή. Είναι η τροπολογία 61. Λέτε ότι η κατασκευή ε, αγαθών μέσω τριδιάστασης εκτύπωσης είναι παράνομη. Δεν μπορεί να έχετε πει παράνομη. Τροπολογία 61. Νομίζω ότι εδώ κάτι έχει γίνει με τη μετάφραση. Ίσως δεν είναι πολύ ακριβής. Θα μου πείτε μετά. Στο, στο τέλος της παρέμβασής μου θα μου πείτε περί τίνος πρόκειται. Ε, γιατί αυτό το παράνομο, δηλαδή ε, κατά του νόμου, κατά της δημοσίας τάξεως, ε, κατά των ηθών, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση τώρα με την αστική ευθύνη, οι τροπολογίες 100 μέχρι 106 ευθυγραμμίζονται όλες, δηλαδή ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η γενική αστική ευθύνη, η οποία θα αφορά και και θα εφαρμόζεται και στην τρισδιάστατη εκτύπωση, ωστόσο μπορούν σε περίπτωση μελλοντικών νομικών επιπλοκών να προκύψουν ε, νέα νομοθετήματα. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ε, ε, αναφερθούμε στη γενική αστική ευθύνη. Ε, φυσικά, τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και ο καθένα έχει τι δικέ του ευαισθησίε. Ε, συμφωνώ απολύτω με την τροπολογία Άντερσον 97 και τη κυρία Χαουτάλα όσον αφορά το ρόλο που θα παίξει η τρισδιάστατη εκτύπωση στην μείωση τη κατανάλωση ενέργεια και φυσικών πόρων, κυρίω όσον αφορά την κατασκευή. Εδώ ο αντίκτυπο μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο και μπορεί η επίπτωση στο περιβάλλον επίσης να είναι πολύ σημαντικός και μπορεί να καταπολεμήσει ακόμα και την κλιματική αλλαγή και επομένως θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσω το σημείο αυτό. Κύριε Γκασμπάρα τροπολογία 111. ανησυχείται για την ποιότητα των προϊόντων που έχουν ε, δημιουργηθεί μέσω της διάστατης εκτύπωσης ε, και ε, συμπληρώνεται λοιπόν την παράγραφό μου 3 και την τροπολογία μου 116 όσον αφορά ε, τα όσα καλύπτονται από την τροπολογία 111. Όσον αφορά τώρα τα πνευματικά δικαιώματα, τα διανοητικά δικαιώματα, καθώς επίσης και τις νομοθετικές και λοιπές τεχνικές ελέγχου, ε, λέτε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα θεσπιστή μάλλον ένας φόρος για την τριδιάσταση εκτύπωσης, εκτύπωση που να καλύπτει τον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τροπολογία 115 Καρή με 118, 119 του κυρίου Γκράντε Γκράντε Πασκουάλ, καθώς επίσης και τροπολογία Μπούντα. Κατανοώ είναι την θέση σας, είναι ένα σημείο αντιφατικό αλλά θα ήθελα να σας εξηγήσω τη θέση μου όσον αφορά ε, την εκτύπωση και τις φωτοτυπίες υπάρχει με ένας ε, φόρος που πληρώνεται όλοι έστω και αν δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι το πληρώνεται είναι 0,001 ε, εκατοστά είναι ανώδυνη αλλά, ο, για τον καθένα αλλά συνολικά είναι ένα σεβαστό ποσό το οποίο τελικά δίνεται στους δημιουργούς. Δεν είναι ένας πραγματικός φόρος, είναι ελάχιστα ψηλά τα οποία μπορούν ε, πραγματικά να κάνουν μια μεγάλη διαφορά για τους δημιουργούς. Ξέρω ότι έχουμε κατακλειστεί όλοι από διάφορους φόρους, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι μια οδός την οποία μπορούμε να διερευνήσουμε, γιατί ε, ε, το συνολικό ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο ε, και δίνεται, αποδίδεται πλήρως στους δημιουργούς ε, και αφορά την ε, εκτύπωση και τα αντίγραφα. Αλλά βεβαίως αν δεν συμφωνείτε με την θέσπιση αυτού του φόρου δεν θα επιμείνω στη θέση μου. Στο iPhone, ας πούμε, τη τελευταίας γενιάς ε, που κοστίζει 800 ευρώ, ε, το 5S. Με αυτό μπορείτε να κάνετε ό,τι φωτογραφίες θέλετε. Υπάρχει ένας φόρος πάνω σε αυτό και μπορείτε και να εκτυπώσετε ό,τι θέλετε. Ε, δεν κοστίζει τίποτα σε σχέση με την αγορά της συσκευή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους δημιουργούς. Συμφωνώ με την κυρία Γκέμπχαρτ όταν λέει ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι απαραίτητη έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και για τα δικαιώματα και την προστασία μάλλον των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία σε σχέση με την τρισδιάσταση εκτύπωση. Πιστεύω δε ότι στο θέμα αυτό τη τρισδιάστασης εκτύπωση εκτύπωσης και την ε, ε, τέχνη δεν έχουμε ακόμα σωστά μετρήσει τον αντίκτυπο αυτής ε, της τρισδιάστασης εκτύπωσης γιατί σε μερικά χρόνια ίσω θα μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα τέχνης που δεν θα μπορούν κανείς να τα ξεχωρίσει από τα πρωτότυπα. Αυτά. Σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ και θα περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις σας και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και από μένα, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Δεγκράντης Πασκουάλ έχει πρώτος το λόγο. Καλημέρα σας κύριε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είχα ήδη την ευκαιρία, όπως και οι υπόλοιποι, να εκφραστούμε πάνω στο θέμα αυτό στην πρώτη ανταλλαγή που είχαμε στην Επιτροπή Νομικών ε, Υποθέσεων. Τώρα βλέπω ότι στις ε, τροπολογίες υπάρχει αρκετά μεγάλη ταυτοσημεία όσον αφορά ε, τις θέσεις που έχουν μέσω των τροπολογικών εκφραστεί. Δεν ε, νομίζω ότι έχουμε έτσι σημαντικά προβλήματα και αντιπαράθεση με την εισηγήτρια την οποία ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητά της και τη γενική στάση που έδειξε. Εγώ έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες τις οποίες με πολύ καλή διάθεση αντιμετώπισε Είναι γεγονός ότι στην αξιολόγηση που κάνουμε ε, έχουμε διαφορετική εκτίμηση όσον αφορά τις νέες δυνατότητες που μπορεί να φέρει αυτή η νέα τεχνολογία για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, οι αξιολογήσεις ε, που κάνουμε δεν είναι ειλικρινείς ε, και ορθές και από τις δύο πλευρές. Εγώ πάντως και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τα πόδια μας στη γη, να είμαστε ε, να μην ε, είμαστε θεροβάμονες στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή εδώ ε, μιλάμε για το αυτόνομο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουμε ακόμα καθορίσει τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητο να λυθούν πριν αρχίσει να λειτουργεί αυτό το νέο μηχάνημα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα γιατί η πραγματικότητα είναι ε, ε, συγκεκριμένη και την πραγματικότητα θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας όταν αναλύουμε αυτά τα θέματα. Βεβαίως ε, <clears throat> τα πλεονεκτήματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης για τις καινοτόμες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικά τους επιτρέπει να μειώσουν το γενικό τους κόστος, να δοκιμάσουν νέα προϊόντα, ε, να βελτιώσουν τα υπάρχοντα προϊόντα κτλ. Ε, μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία μπορεί ε, να κάνει πιο προσιτά ορισμένα αντικείμενα τεχνολογία σε όλο τον κόσμο και να διευκολύνει εν τέλει τη ζωή μας με πολλούς ε, βουλευτές ε, που δεν θα ονομάσω, αλλά είναι η πλειοψηφία, ε, έχουμε υποβάλει τροπολογίες οι οποίες είναι, πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Τις ανέφερε η κυρία εισηγήτρια αναλυτικά τις τροπολογίες αυτές και μάλιστα ανέφερε τροπολογίες οι οποίες οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση και εγώ θέλω να το τονίσω αυτό γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό προερχόμενες οι τροπολογίες αυτές κυρίως από διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Τέλος, να πω ότι έχουμε διαφορά όσον αφορά την θέσπιση φόρου για την τρισδιάσταση ε, εκτύπωσης. Υπάρχουν ήδη τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Εγώ δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω. Είσαστε όλοι ε, νομικοί και νομομαθείς ε, ε, επομένως, σας λέω ότι η θέση μου απέναντι σε ένα νέο φόρο δεν είναι πάντα η ίδια. Ε, ούτως ή άλλως, εδώ μιλάμε για καθαρά εθνικές αρμοδιότητες και εδώ νομίζω ότι παρεμβαίνουμε και ξεπερνάμε τα όρια της επικουρικότητας προτείνοντας κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε υποβάλει 24 τροπολογίες ε, ε, επί συνόλου 149 τροπολογιών, όπως μας έλεγε ε, η συγγήτρια. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν θέσεις οι οποίες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να βρουν κοινό τόπο. Αντιθέτως, Πιστεύω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε τα κριτήρια ε, που έχουν ακολουθήσει οι διάφοροι υποβάλλοντες τροπολογίες. Ε, μπορούμε να ακολουθήσουμε και τη λογική ε, της εισηγήτριας έτσι ώστε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή σε τούτη την έκθεση. Τελειώνοντας να συγχαρώ την εισηγήτρια και για την εργασία της αλλά και για τη γενική της στάση και ευελπιστώ ότι όσο γίνεται πιο πολύ θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα θέματα τα οποία τίθενται μέσω των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους ε, της ε, κυρίας Δελβού, της ε, Σκιώδους από το S.N.D. η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα. Και για τους διερμηνείς τώρα θα γυρίσω στα γαλλικά Έχοντας διαβάσει πολύ προσεκτικά την έκθεση της κυρίας Μπερζερόν, συμφωνώ με την πρωτοβουλία της, υπέβαλε τροπολογίες όμως για πάρα πολλά σημεία. Όσον αφορά τα εκτιμώντα, την τολική σκέψη δηλαδή, θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε ένα κείμενο το οποίο βρίσκεται ακόμα υποσυζήτηση. Αναφορά στα άρθρα 10 και 14, καθώς επίσης και σε προτάσεις που γίνονται όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου θα προτιμούσε να γνώριζε το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών προτού προβλεφθεί η εφαρμογή του. Η κυρία Μπερζερό αναφέρθηκε στο σημείο αυτό και νομίζω ότι όντω είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε για το τι ακριβώ μιλάμε εδώ πέρα και το κείμενο ακόμα δεν έχει παγιωθεί. Όσον αφορά το ζήτημα της ευθύνη για την ανάπτυξη τρισδιάστατης εκτύπωσης σε βιομηχανική κλίμακα, θεωρεί ότι θα πρέπει εδώ πέρα να υπάρχει δυνατότητα συλλογική προσφυγής, προκειμένου να αποζημιώνονται οι ζημιωμένοι καταναλωτές. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στο εκτιμώντας M10 με τον ίδιο στόχο προστασία, δηλαδή των καταναλωτών, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα ταυτοποίηση και εντοπισμού, προκειμένου να υπάρχει πραγματικά η χτυλασιμότητα των προϊόντων και αναφερόμαστε εδώ πέρα στην παράγραφο 3. Υπενθυμίζει ότι η νέα αυτή τεχνολογία έχει πολλά οικονομικά προνόμια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω για τη δυνατότητα εξατομίκευση κάποιων προϊόντων και αυτό όντω αντιστοιχεί σε κάποια, σε κάποια αποτετήματα των Ευρωπαίων καταναλωτών. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται επίση εξοικονόμηση ενέργεια και δεν υπάρχει το απαραίτητο συντεκτικό τοπικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει μια εναρμονική μετάβαση στον νέο αυτό Η κυρία Ντελβό είναι αρκετά διαλλακτική για να βρεθούν συμβαστικές λύσεις και να γίνουν περισσότερες συζητήσεις. Θα ήθελα τώρα να σας πω όσον αφορά ε, την ε, ε, τροπολογία 123 η οποία είπατε ότι είναι θετική. Έχω ένα πολύ σημαντικό ερώτημα διότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να έχει θετικές συνέπειες όμως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τι σημαίνει και για την αναπαραγωγή και τα δικαιώματα των συγγραφέων και πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το ερώτημα ερώτημα ε, και ε, με ένα ε, με μια επιπλέον πληρωμή δεν θα επιληθεί. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ώστε σε αυτούς τομείς να αναλογιστούμε και τα δικαιώματα των συγγραφέων. Ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την συγγήτρια για το έργο της ε, και θα πω κάτι εντάχει. Έχω ε, καταθέσει 23 τροπολογίες, δεν θα τις αναφέρω όλες, όμως ε, ε περιληπτικά θα ήθελα να πω ότι η νομοθέτηση της τριδιάστατης εκτύπωσης ε, θα πρέπει να το ε, διευκολύνει ούτω ώστε να αναπτυχθεί και η κοινωνία να μπορέσει να ε, χρησιμοποιήσει αυτήν την υπέροχη νέα τεχνολογία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε πολλή νομοθεσία ή κακή νομοθεσία η οποία θα θέσει εμπόδια σε αυτή την τεχνολογία. Όσον αφορά την τροπολογία 61 στην αιτιολογική σκέψη, σκέψη H ενημερώθηκα από τη γραμματεία ότι υπήρξε λάθος μετάφραση στα γαλλικά, αν καταλαβαίνω λοιπόν ορθά και συγγνώμη ε, για την προφορά μου. Νομίζω ότι λείπει μία λέξη. Ε, ακούγεται πολύ καλύτερα, ε, βγάζει περισσότερο νόημα ε, στα αγγλικά και αφορά την αλλαγή της αιτιολογικής σκέψης H ε, που ε, δεν βγάζει πολύ νόημα ε, στα αγγλικά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα καταρθώσουμε να έχουμε μια συμφωνία πάνω σε αυτήν την αιτιολογική σκέψη. Τώρα όσον αφορά την τροπολογία την παράγραφο 4 η τροπολογία μου 116 αφορά ε, την αφαίρεση της φορολόγησης της τρισδιάστητης ε, τεχνολογίας ε, διότι θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Δεν βλέπουμε λοιπόν κάποιο συσχετισμό μεταξύ των διαφόρων φόρων που έχουμε στις φωτοτυπίες, στα κινητά τηλέφωνα όταν έχουν ένα, ένα αρχείο. Όταν όταν ε, λοιπόν αγοράζεις ένα αρχείο από τρισδιάστατο εκτυπωτή, ο πρωταρχικός ε, σκοπός αγοράς ενός τέτοιου, ε, ενός τέτοιου αρχείου είναι να χρησιμοποιηθεί. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να υπάρχει ένας φόρος φωτοτυπίας. Όσον αφορά την παράγραφο 5, ε, ε, η τροπολογία 125 αφορά την αφαίρεση της παραγράφου 5, διότι ανησυχούμε για, το, ε, για τα για την υπερβολική παρακολούθηση που δημιουργείται. Επίσης ε, πιστεύουμε ότι η οδηγία για το, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ε, καλός, ε, θα πρέπει να ε, γίνει σεβαστός. Έχουμε ε, διάφορες τροπολογίες για αυτό το θέμα, όπως είναι για παράδειγμα η τροπολογία 141 ε, που αφορά την εφαρμοσιμότητα ε, των συγκεκριμένων αρχείων ε, θεωρεί κατάλληλε τι υποδομέ υπηρεσιών ε, τρισδιάσταση εκτύπωση, οπότε πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό. Η κυρία Μπουτόντα έχει το λόγο. Το μικροφόνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπερζέρο για την έκθεσή της και τις εξηγήσει που έδωσε. Όπως υπόθηκε όντω, έχω καταθέσει και εγώ αρκετές τροπολογίες. Συμφωνώ με τη διαπίστωση που γίνεται ότι οι νομικοί κανόνες θα πρέπει να πλαισιώνουν την ε, τεχνολογία και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελούν τροχοπέδι. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας φόρος για τα ιδιωτικά αντίγραφα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό για τους δημιουργούς. Η καινοτομία αυτή πάντω τη τρισδιάστατη εκτύπωση δεν έχει αναστατώσει το εφιστάμενο καθεστώ δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησία και δικαιωμάτων του δημιουργού. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό τα προϊόντα τα οποία θα προκύψουν από την τρισδιάστατη εκτύπωση να μπορούν να χαίρονται μια κάποια προστασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο τα προϊόντα αυτά, δημιουργώντα το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Έτσι προωθούμε και τη τρισδιάστατη εκτύπωση ω τεχνολογία. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα θέλαμε να χαιρετήσουμε το σχέδιο αυτό έκθεσης, το οποίο θέτει κάποια σημαντικά ζητήματα. Θα περιοριστώ στο ζήτημα εκείνο που έχει να κάνει με την αστική ευθύνη και θα ήθελα να σας δώσω κάποιες περαιτέρω πληροφορίες επ' αυτού. Στις 9 Μαρτίου, οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησαν μία πρόσκληση ε, συμμετοχή υποψηφιωτήτων εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ζήτημα τη αστική ευθύνη όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση. Θα ασχοληθεί η ομάδα αυτή εμπειρογνωμόνων με την οδηγία όσον αφορά την ε, ευθύνη, την αστική, και μια άλλη ομάδα θα εξετάσει το ζήτημα από μια πιο ευρία οπτική γωνία. Θέλουμε λοιπόν και εμεί να ασχοληθούμε με τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την αστική ευθύνη, γιατί συνδέονται και αυτά με την ασφάλεια δικαίου, που είναι ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω εξέλιξη αυτή τη νέα καινοτόμα τεχνολογία υπέρ των πολιτών, υπέρ των καταναλωτών. Η 30 Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να υποβληθούν υποψηφιότητε για αυτήν την ομάδα πυρογνωμόνων. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Δεν ξέρω αν η κυρία τώρα θα ξαναπάρει το λόγο. Πολύ απλά και να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Δεγκράντερ Πασκουάλ. Ο κύριος Δεγκράντερ Πασκουάλ όντω έκανε κάποιε πολύ θετικέ παρατηρήσει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προστατεύουμε το καταναλωτή και το περιβάλλον, χωρί όμω να αναχαιτήσουμε το ρυθμό εξέλιξη αυτή τη νέα τεχνολογία. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε στον νέα αυτή τεχνολογία. Λαμβάνω υπόψη τα όσα είπατε. Βλέπω ότι υπάρχει μια διάσταση απόψε όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού. Εγώ λόγω τη ε, κατάρτιση που είχα και των σπουδών που έχω κάνει θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προστατεύσουμε του δημιουργού χωρί του δημιουργού δεν θα υπήρχε ουσιαστικά και πολιτισμό. Η τρισδιάστατη λοιπόν εκτύπωση αποτελεί καταπληκτική ευκαιρία πολύ συχνά και για όσου παραποιούνται τα διάφορα προϊόντα για τους α, όσους προχωρούνται σε παραχαρά, παραχάραξη των προϊόντων αυτών. Όταν για παράδειγμα δημιουργείται τα κόσμημα, το οποίο δημιουργεί ο οικοσκαρτιά για παράδειγμα, ξέρετε ότι προβλέπετε μια ολόκληρη εργασία από πίσω. Αν εσείς συνεχεία μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορείτε να αναπαράγετε το ίδιο αυτό κόσμημα καταλαβαίνετε ότι η υπογραφή πλέον του οίκου, ο Δημιουργό, και ουσιαστικά τα δικαιώματα που τα αντιστοιχούνται δεν θα ισχύονται πλέον, γιατί μπορείτε εσά να δημιουργείτε εκ νέου το προϊόν αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προστατεύσουμε τον ίδιο τον δημιουργό, την ίδια τη δημιουργία, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τον ίδιο τον πολιτισμό μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξαναπώ ότι... Ε, στις 24 Απριλίου προβλέπεται να ε, γίνει το θέμα, να συζητηθεί στην ε, στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, έχουμε τώρα την, τη συμβάση σε παροχή ψηφιακού περιεχομένου. Θα δώσω ξανά το λόγο στο σημείο 6. Είμαστε στην κυρία Ευλίν Κέμπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πιστεύω ότι ε, διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στην ε, Βουλγαρική Προεδρία για την ε, προσπάθεια που κάνει να πείσει τα, τα, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ούτως ώστε να έχουμε έναν καλό συμβιβασμό. Ε, έχουν γίνει πρόοδοι από την τελευταία συνεδρίαση, ιδιαίτερως όσον αφορά την αξία των updates και ε, για πόσο καιρό θα πρέπει να ισχύουν. Ε, είναι ένα από τα σημεία οποία, στα οποία διαφωνούσαμε και πιστεύουμε ότι οι κανονισμοί που βρήκαμε θα έχουν αισιόδοξα αποτελέσματα, διότι κάνουν μια διαφοροποίηση μεταξύ των updates για την ασφάλεια που είναι πολύ σημαντικά και περαιτέρω περαιτέρω ε, updates, ε, τα οποία επίσης είναι σημαντικά, ε, αλλά έχουν διαφορετική αξία σε σχέση με την ασφάλεια των ανθρώπων. Ένας άλλος τομέας στον οποίο έχουμε συμφωνήσει αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε το δίκαιο προστασίας δεδομένων, ιδιαιτέρως την, το, τον κανονισμό, το γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων είπαμε και το έχουμε εφαρμόσει ότι ως κοινοβούλιο και στο κείμενο το οποίο θα ε, καταρτήσουμε ότι όσον αφορά ε, παραβιάσεις του γενικού κανονισμού ε, θα λαμβάνονται και τα κριτήρια συμβιβασμού αλλά θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά ε, αφορά ε, τα, ε, τα ενσωματωμένα ψηφιακά περιεχόμενα, αν θα πρέπει αυτά να συμπεριλαμβάνονται ή όπως πρότεινε η Κομισιόν να, συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στον κανονισμό γενικών προϊόντων. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διαφορετικό δίκαιο για μια προεγκατεστημένη εφαρμογή σε κάποιο κινητό ε, και ε, μια ένας διαφορετικός κανονισμός για το update του. Ε, θα πρέπει, αν υπάρχει διαφορετικό δίκαιο, τότε ούτε ο καταναλωτής, ούτε ο πολιτής ή η επιχείρηση θα μπορούν να διακρίνουν τι είναι τι και γι' αυτό το λόγο εμένουμε ότι ε, το ε, ψηφιακό ε, περιεχόμενο, όχι το ίδιο το κινητό, αλλά οι εφαρμογές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και εκεί χρειαζόμαστε λοιπόν λίγο έργο ακόμα. Ε, δεν έχουμε ε, πάντοτε την συμφωνία της Κομισιόν, ε, όμως είναι ένα σημαντικό θέμα για εμάς. Ένα άλλο σημείο τώρα, στο οποίο δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα, αφορά το επίπεδο εναρμόνισης. Το Κοινοβούλιο θέλει πλήρη εναρμόνιση, το οποίο είναι και λογικό διότι ε, πέραν των κάτω χωρών και, της, ε, και του Ηνωμένου Βασιλείου ε, δεν υπάρχει νομοθεσία στα άλλα κράτη-μέλη συγκεκριμένη για αυτό. Έτσι λοιπόν κάποιοι θέλουν την ελάχιστη εναρμόνιση, άλλοι όχι. Είναι, κάποια, είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, όμως... η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι θετική μέχρι ε, στιγμής Και έτσι λοιπόν βλέπω, έχω την εντύπωση, την ότι ε, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας ε, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά βέβαια, βλέπω όμως ότι υπάρχει ε, μια ευκαιρία εδώ πέρα. Ε, έχουν μείνει μονάχα δύο σημεία, όλα τα άλλα μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει βούληση και από τις ε, δύο πλευρές να υπάρξει γρήγορα ένας ε, κανονισμός για έναν τομέα ο οποίος εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με τα ενσωματωμένα ψηφιακά περιεχόμενα. Βλέπουμε ε, λοιπόν ότι ε, η πρόταση για τα ενσώματα αγαθά ε, είναι ίσως το μέλλον και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο διότι για παράδειγμα πρόσφατα αγόρασα έναν καινούριο ποτή τον εγκατέστασα και συνειδητοποίησα ε, ότι ε, μπορώ να το συνδέσω ε, και με τον υπολογιστή όμως δεν το έκανα διότι δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχει κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς καμία ρύθμιση διότι είναι τομείς που είναι σημαντική για τους πολίτες και η ασφάλεια σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντικό έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση. Ελπίζω να σας έχω, να σας έχω ενημερώσει καλά και παραμένω στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ ε, για τα καλά νέα. Θα ήθελε κάποιος άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται η Κομισιόν, μήπως έχει να μας πει κάτι. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η εντύπωσή μας από πλευράς Κομισιόν είναι ταυτόσιμη με αυτή που εξέφρασε μόλις η κυρία Γκέπχαρτ. Ε, έχει ήδη γίνει ικανή πρόοδος και ε, πιστεύουμε ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πολιτική συμφωνία υπό την Βουλγαρική Προεδρία. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε ε, την εργασία έρχοντας αυτόν τον στόχο. Ίσως θα μπορούσα να πω ε, για το θέμα του ενσωματωμένου ψηφιακού περιεχομένου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πριν από λίγο συζητούσαμε την τρισδιάστατη εκτύπωση. Ε, όλο και περισσότερα προϊόντα στο μέλλον θα είναι ψηφιοποιημένα και επομένως χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια και, σαφήνη, και βεβαιότητα για τα θέματα αυτά. Είναι πολύ ευαίσθητα και δείχνουμε και εμείς την ίδια ευαισθησία για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Τώρα δουλεύουμε σε ένα paper που ζητήθηκε από την Κομισιόν έτσι να δούμε ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι ορθοί κανόνες ε, για την αντιμετώπιση αυτού του ενσωματωμένου ψηφιακού ε, περιεχομένου. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τα κατάλληλα εργαλεία, μετά να δούμε σε ποιο ε, μηχανισμό ή εργαλείο θα πρέπει να ενσωματωθούν, γιατί το σημαντικό είναι οι κανόνες που θα προκύψουν να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά για το καλό των καταναλωτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν φαίνεται να ζητά κάποιο άλλο το λόγο, Επομένω μπορούμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό και να φτάσουμε στο σημείο 7. Είναι η αναφορά σχετικά με την πρόοδο των διαδικασιών και διαπραγματεύσεων όσον αφορά ε, θέματα ε, για τα οποία εγώ ήμουν επικεφαλής. Ε, δεύτερος πρόεδρο, δεύτερη, δεύτερος τριμερής διάλογος ως όσον αφορά τα τηλεοπτικά προγράμματα κτλ. Εγώ ήρθα σε επαφή με την κυρία Κούλεβα, με την κυρία Γκαμπριέλα από πλευρά τη Κομισιόν. Ε, κάναμε πρόοδο σε σχέση με κάποια θέματα τα οποία προετοιμάστηκαν ε, σε τεχνικό επίπεδο πριν από τον τριμερή διάλογο. Δυστυχώς όμως δεν έγινε πολύ σημαντικός ουσιαστικός διάλογος όσον αφορά τα τέσσερα ζητήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί ως κύρια πολιτικά ζητήματα στον πρώτο τριμερή στο μεγαλύτερο μέρος του τριμερούς ε, διαλόγου αποσαφηνίστηκαν οι θέσεις των τριών ε, ε, οργάνων όσον αφορά θέματα που αφορούν το εύρος, την αναμετάδοση, την άμεση παρεμβολή καθώς επίσης και την ημερομηνία εφαρμογής. Εργαζόμαστε τώρα σε τεχνικό επίπεδο ε, και ο τρίτος ε, τριμερής ε, διάλογος θα λάβει χώρα την 17η Απριλίου στο Στρασβούργο. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω εγώ. Δεν ξέρω εάν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο, από ό,τι φαίνεται όχι. Και επομένως μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη και του θέματος αυτού και να φτάσουμε στο σημείο υπαριθμών 8. Αφορά το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας δυνάμει του κανονισμού 726 κάθετος 2004 για ένα ορφανό φάρμακο η ε, εισηγητής είναι ο κύριος Γιένς Ρόντε, ο οποίος μου ζήτησε να σας πω ότι δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτήν την εκτελεστική απόφαση. Έχει κάποιος άλλος διαφορετική απο... Ε, άποψη? Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένως ολοκληρώνουμε και την εξέταση του σημείου 8 και περνάμε στο σημείο 9 το οποίο αφορά μελέτη σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας που χορηγήθηκε βάσει της απόφασης C 2014 ε, τελικό 5318 τελικό όσον αφορά επίσης ένα φάρμακο ε, ο εισηγητή είναι πάλι ο κύριος Γιάννης Ρόντε, ο οποίος ε, επαναλαμβάνω ότι και για την προκείμενη περίπτωση ε, δεν έχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά την υιοθέτηση αυτή της εκτελεστικής απόφασης. Δεν ξέρω εάν κάποιος συνάδελφος έχει άλλη αντίθετη γνώμη. Όχι, ολοκληρώθηκε το θέμα 9 και περνάμε στο σημείο 10. Uh, Σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 1352 του 2013, η συγητής για μία ακόμα φορά είναι ο κύριος Ρόντε και για μία ακόμα φορά σας επαναλαμβάνω τον εκπρόσωπο και ότι δεν έχει καμία ε, ε, πρόθεση αντίθεσης όσον αφορά αυτήν την τροποποίηση και αυτόν τον εκτελεστικό κανονισμό. Περνάμε επομένως απευθείας στο σημείο 11. που αφορά εξέταση κατεξουσιοδότηση κανονισμού της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 217 κάθετος 1001 ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση του κατεξουσιοδότηση κανονισμού 2017 κάθετος 1430. Εισηγητής είναι ο κύριος Γιένς Ρόντε. Για μία ακόμα φορά μου ζήτησε να σας πω ότι δεν βλέπει καμία, κανένα λόγο να αντιταχθεί σε αυτήν την ε, διαδικασία. Στις 23 ε, Μαρτίου Παρασκευή έλαβα ε, επιστολή ε, από την Επίτροπο Μπινκόφσκα όπου μου ζητά ακριβώς να μην ενταχθούμε σε αυτήν την κατεξουσιοδότηση πράξη. Χθες κυκλοφόρησε επίσης και μία επιστολή ε, προς τον πρόεδρο της CCC ε, σύμφωνα και με τον κανονισμό 105 εδάφιο 5 του κανονισμού λειτουργίας. Ε, σε αυτήν την περίπτωση και αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση ε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σε επίπεδο επιτροπής. Η Γραμματεία θα αναλάβει ε, όλες τις τεχνικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υποβληθεί εις την Ολομέλεια το, το αντίστοιχο νομοθετικό ψήφισμα το οποίο θα δοθεί μετά στην κυρία Βίκστρομ αυτά σχετικά με το θέμα αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε. Σημείο 12 το οποίο αφορά την επικουρικότητα, αυτό είναι μόνο προσημείωση. Και επομένως τώρα θα πρέπει να σταματήσουμε γιατί είμαστε εξαιρετικά αποτελεσματικοί, ταχύτατοι και η ψηφοφορία έχει προβλεφθεί για τις 11. Επομένως δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σε μία ώρα θα τα πούμε λοιπόν. Διακόπτουμε. Α, ο κύριε Χρυσόγονε, παρακαλώ. Κύριε Χρυσόγωνε, ο κύριος Χρυσόγωνε θέλει το λόγο. Εάν θέλετε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το θέμα 22 τώρα που αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής ε, του Ευρωπαϊκού Νόμου για το 2013. Εγώ στρέφομαι προς ε, τα μέλη. Θέλετε να το κάνουμε αυτό? Θέλετε δηλαδή να εξετάσουμε το θέμα 22 του κυρίου Χρυσόγονου. Η απάντηση από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι θετική και επομένως, και επομένως μπορούμε να ε, πάμε στο θέμα 22, το οποίο αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 και δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Χρυσόγων. So, uh... Thank you, uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την εκδομοσύνη μου προς τους συναδέλφους από την Επιτροπή για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Και θα ήθελα να τονίσω ότι περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές είναι τροπολογίες οι οποίες μπορώ να δεχτώ. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες αυτές όντως βελτιώνουν το κείμενο το οποίο προετοίμασα και προτίθεμαι αποδεκτώ τις περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες. Σε κάθε περίπτωση, τα βασικά ζητήματα τα οποία έθεσα στα πλαίσια της έκθεσής μου και για τα προηγούμενα έτη, εξακολουθούν να υφίστανται και για το έτος 2016, όσον αφορά τα την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε αν όχι ομοφωνία, τουλάχιστον μια ευρεία συνένεση για τα ζητήματα αυτά, όπως ακριβώς είχαμε κάνει και με τις ανάλογες εκθέσεις για τα προηγούμενα έτη. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε κύριε Χρυσόγοντα. Υπάρχει κάποιος που θα θέλει να πάρει το λόγο. Το σχέδιο έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως ούτε και αυτή. Δεν έχω παρά να σας ενημερώσω ότι προβλέπεται να ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή στην Επιτροπή μας στις 23 και 24 Απριλίου. Άρα κλείνουμε και το σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης και δεν μπορούμε να αποφύγουμε το διάλειμμα μας μέχρι τις 11.